Okay, colleagues. Um, Αγαπητοί συνάδελφοι, είχαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα ανταλλαγή απόψεων σήμερα το πρωί, αλλά εξίσου ενδιαφέρονταν και τα υπόλοιπα σημεία στην ημερήσια διάταξη. Το πρώτο έχει να κάνει με την εφαρμογή τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία. Ζήτημα πάρα πολύ σημαντικό και για τη δική μα την Επιτροπή, πριν από μερικές μέρες άκουσα ένα πρόγραμμα στο ραδιόφωνο σχετικά με την ε, νομοθεσία του Ηνωμένου Βασιλείου όσον αφορά τα άτομα με αναπηρίες. Πριν από λίγο καιρό, το 1985, ένας νέος ήθελε να πάει στον κινηματογράφο, ήταν ανάπηρος, δεν μπορούσε να πάει σε κανένα κινηματογράφο στη Βρετανία, δεν τον άφηνα να μπει μέσα γιατί υπήρχε κίνδυνος για πυρκαγιά και δεν θα μπορούσε ενδεχομένω να αποχωρήσει εύκολα από την αίθουσα. Θεωρώ ότι και στη Μεγάλη Βρετανία αλλά και σε πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος όσον αφορά τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία. Τα δικαιώματα αυτά θεωρούνται πλέον θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα. Υπάρχουν όμως και άλλες πλευρές του κόσμου, άλλες περιοχές του κόσμου όπου η πρόοδος αυτή δεν έχει ακόμα επιτευχθεί. Υπάρχουν χώρες που έχουν μεγάλους αριθμούς ανθρώπων με αναπηρία, οι οποίες θα πρέπει να σημειώσουν πολύ πιο σημαντική πρόοδο από αυτή που έχουν σημειώσει μέχρι στιγμή. Χαίρομαι πάρα πολύ που μαζί μα τον Λάρς Μπόσελμαν, ο οποίο είναι διευθυντή του Διεθνού Κονσόρσιου ανάπτυξη και Ατόμων με Αναπηρία. Ασχολείται λοιπόν με τη διασύνδεση ανάμεσα στι πολιτικέ για την αντιμετώπιση της αναπηρία ή την πρόθεση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία και τις πολιτικές ανάπτυξης στα πλαίσια της Ατζένα 2030. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να καλημερίσω και όλα τα μέλη της Επιτροπής σας. Να σας πω καταρχάς ποια είναι η δική μου η οργάνωση. Συμμετέχουμε στο Διεθνές Κονσόρσιουμ για την Ανάπτυξη και τα άτομα αναπηρία. Εγώ εργάζομαι όμως συγκεκριμένα για το CBM, που είναι ένας οργανισμός για την πρόθεση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία σε χώρες μεσαίου και χαμηλού εισοδήματος. Ενδεχομένω να είναι ιδιαίτερα ευρία η εντολή μου, εκ πρώτη όψεω τουλάχιστον, καλύπτουμε όντω πάρα πολλού τομεί, όπω τον τομέα τη εκπαίδευση, τη υγειονομική περίθαλψη, αλλά και προσπαθούμε επίση να υποστηρίξουμε εν γέννη το κίνημα πρόθεση των δικαιωμάτων των ατόμων με σε διάφορε αναπτυσσόμενε χώρε. Μέρος της εργασίας μου είναι και μια εργασία πολιτικής φύσης που περιλαμβάνει τελικά τη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με άλλους δωρητές, αλλά επίσης και με υπηρεσίες των Ηνωμένων Εθνών, προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία βρίσκονται στις πρώτες θέσεις ε, της πολιτικής ατζέντα όλων αυτών των οργανισμών. Σε επίπεδο Ηνωμένων Εθνών γίνεται μια σημαντική εργασία, αλλά συνεργάζομαι και με άλλους οργανισμούς όπως η Concord, την οποία τη γνωρίζετε προφανώς όλοι. Ελάχιστο είναι ο χρόνο που έχω στη διάθεσή μου. Θα πρέπει λοιπόν να επικεντρωθώ πολύ σύντομα σε πολύ συγκεκριμένα σημεία. Θα μπορούσα να μιλάω πάρα, πάρα πολύ ώρα για το πολύ σημαντικό και ενδιαφέρον αυτό ζήτημα. Παρ' όλα αυτά θα ήθελα να επικεντρωθώ σε δύο συγκεκριμένα σημεία. Πρώτον, να περιγράψω λίγο καλύτερα κάποιες βασικές πτυχές της ε, παγκόσμιας κατάστασης των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία σε αναπτυσσόμενες κυρίως χώρες. Αυτό μας ενδιαφέρει εμπροκειμένο και από την άλλη θα ήθελα να κάνω και κάποιες συγκεκριμένε ε, προτάσεις ε, για το πώς μπορούμε να ενισχύσουμε το κείμενο της γνωμοδότησης το οποίο θα σας παρουσιάσει η κυρία Χάουταλα μετά τη δική μου την παρέμβαση, κείμενο το οποίο το έχετε λάβει όλοι σας. σε παγκόσμιο επίπεδο τι συμβαίνει με τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία. Θα έλεγα ότι καταρχάς θα πρέπει να σκεφτούμε εδώ πέρα ότι αναφερόμαστε σε πολύ σημαντικούς αριθμούς. Ένα περίπου 15% του παγκόσμιου πληθυσμού ζει με μία μορφή τουλάχιστον αναπηρίας και από τους ανθρώπους αυτούς περίπου το 80% ζουν σε αναπτυσσόμενες χώρες. Αυτό από μόνο του μας δείχνει από ποσοτικής πλευράς πόσο σημαντικό είναι το ζήτημα. Το φαινόμενο αυτό επηρεάζει πάρα πολλούς ανθρώπους σε αναπτυσσόμενες κυρίως χώρες, αλλά προφανώς και σε αναπτυγμένες χώρες. Η δεύτερη πτυχή της παγκόσμιας αυτής εικόνας που θέλω να σας δώσω είναι ότι η αναπηρία είναι αιτία αλλά και συνέπεια της ένδυας και της φτώχειας. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που ζουν με αναπηρίες σε φτωχές χώρες, σε φτωχές περιοχές οι οποίοι αν είχαν γεννηθεί σε πλουσιότερες περιοχές του κόσμου, ενδεχομένω να μην είχαν καν αυτή την αναπηρία. Και ενδεχομένω αυτό να οφείλεται σε συστήματα υγειονομική περίθαλψης, στην έλλειψη υγειονομικών υπηρεσιών και το καθεξής. Πολύ συχνά όμως έχει να κάνει μόνο με τον υποσυτισμό ή γενικότερα την κακή διατροφή, φαινόμενο το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε αναπηρία. Το γεγονός τώρα ότι οι άνθρωποι ζουν με αναπηρίες από μόνο του τους δίνει λιγότερες ευκαιρίες να καταφέρουν να βγουν από τη φτώχεια. Και αυτή την πτυχή νομίζω ότι θα πρέπει να την καταλάβουμε γιατί είναι πάρα πολύ σημαντική. Πώς γενικά κανείς μπορεί να ξεφύγει από τη φτώχεια. Αυτό έχει να κάνει κυρίως με την εκπαίδευση, με τη δυνατότητα οι άνθρωποι να βρουν μια απασχόληση με σωστά εισοδήματα, με τη δυνατότητά τους να συμμετέχουν σε προγράμματα κατάρτισης και γενικότερα με τη γενικότερη δυνατότητά τους να συμμετέχουν στα κοινά. Καταλαβαίνετε ότι ένα άτομο με αναπηρία σε όλους αυτούς τους τομείς, σε όλες αυτές τις δραστηριότητες, αντιμετωπίζει πάρα πολλούς φραγμούς, πάρα πολλά εμπόδια, τα οποία δεν μπορώ να σας περιγράψω αυτή τη στιγμή με κάθε λεπτομέρεια, αλλά τα περισσότερα έχουν να κάνουν καταρχάς με το υλικό περιβάλλον στο οποίο κινείται ο άνθρωπος αυτός, ενώ άλλα φράγματα, άλλα εμπόδια μάλλον έχουν να κάνουν περισσότερο με την οτροπία της προκαταλήψης που υπάρχουν σε διάφορες χώρες, με τα στερεότυπα, πολλές φορές ακόμα και με την επικρατούσα θρησκευτική πίστη σε μία χώρα ή μόνο και μόνο με το ότι ορισμένες περιοχές ή χώρες δεν έχουν τους απαραίτητους πόρους προκειμένου να παράσχουν στους ανθρώπους αυτούς τις κατάλληλες υπηρεσίες που θα τους βοηθούσαν να βγούνε από το καθεστώς στόχιας. Μία τρίτη πτυχή που πρέπει να δούμε όσον αφορά την παγκόσμια αυτή σφαιρική εικόνα για, τη δικαιώμα, για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία είναι ότι υπάρχουν όλο και περισσότερο επιστημονικά δεδομένα που μας δείχνουν ότι το ότι αποκλείονται τα άτομα με αναπηρία δεν είναι μόνο καταστροφικό για τα ίδια τα άτομα, αλλά είναι καταστροφικό και για την ίδια τη χώρα ή και για την οικονομία της χώρας στην οποία ζουν οι άνθρωποι αυτοί. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό και πρέπει να το καταλάβουμε και είναι κάτι το οποίο να δίεται όλο και περισσότερο σε έβριμα των μελετών που γίνονται σε αυτό το τομέα. Δηλαδή, πόσο πολύ τελικά ζημιώνονται οι ίδιες οι χώρες, οι ίδιες οι κοινωνίες μας όταν αποκλείουν και παραμερίζουν τους ανθρώπους με αναπηρία ενώ θα μπορούσαν τους ανθρώπους αυτούς να τους προσελκύσουν περισσότερο προς προγράμματα κατάρτισης, προς μια πιο αποτελεσματική απασχόληση κ.ο.κ. Και κάτι ακόμα. Πριν από δέκα χρόνια πιστεύω ότι δεν θα συζητούσαμε καν το ζήτημα αυτό. Με άλλα λόγια, η εναπηρία στον απτυγμένο τουλάχιστον κόσμο είναι ένα ζήτημα το οποίο κεντρίζει όλο και περισσότερο τον ενδιαφέρον σε παγκόσμιο και ευρωπαϊκό επίπεδο. Και αυτό από μόνο του είναι μια θετική εξέλιξη. Αρκεί να δούμε κάποια από τα διεθνή πλαίσια, τις διεθνείς συμφωνίες που εγκρίθηκαν πρόσφατα και βλέπουμε ήδη ότι στους στόχους για τη βιώσιμη ανάπτυξη με ορίζοντα το 2030, στους στόχους δηλαδή των ΗΕ, Εθνών, γίνεται ρητή αναφορά στην πρόθεση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία. Τα δικαιώματα όμως αυτά προωθούνται βέβαια και από την ίδια την Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, την CRPD, η οποία υιοθετήθηκε πριν από 10 χρόνια Ξέρετε ότι φέτος γιορτάζουμε την δεκαετή επέτειο της συμφωνίας αυτής και η σύμβαση αυτή των Ηνωμένων Εθνών ασχολείται με το ζήτημα των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία και προσπαθεί ουσιαστικά να μην δημιουργήσει νέα δικαιώματα για τους ανθρώπους αυτούς, αλλά να έχουν όλοι οι άνθρωποι αναπηρία πρόσβαση σε όλα τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση κατάφερε να υπογράψει τη σύμβαση αυτή ως διεθνής φορέας και όχι μεμονωμένα μέσω των κρατών μελών της, αυτό από μόνο του είναι πάρα πολύ σημαντικό και ουσιαστικά η σύμβαση αυτή έχει δύο συγκεκριμένα άρθρα που έχουν να κάνουν με την ανθρωπιστική βοήθεια και την αναπτυξιακή συνεργασία. Δεν θέλω να σας δώσω αυτή τη στιγμή συγκεκριμένους αριθμούς, είναι το άρθρο 11 και το άρθρο 32. Εν συντομία, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχοντας επικυρώσει τη σύμβαση αυτή, υποχρεούται πλέον να ευθυγραμμίσει την ανθρωπιστική της πολιτική και την πολιτική αναπτυξιακής βοήθειας με τη σύμβαση αυτή και θα πρέπει να προωθήσει στους τομείς αυτούς τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία. Από την άλλη, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να διασφαλίσει ότι δεν θα δημιουργεί νέα εμπόδια μέσω των νέων αυτών δραστηριότητών της. Ένα παράδειγμα που θα μπορούσα να σας δώσω για παράδειγμα είναι ότι νέα σχολεία για παράδειγμα τα οποία οικοδομούνται μετά από έναν σεισμό δεν θα πρέπει να εμπεριέχουν νέα εμπόδια ή φραγμούς για τους ανθρώπους με αναπηρία. Θα πρέπει εξ αρχής δηλαδή, κάθε φορά που εκπονείται μια νέα πολιτική, κάθε φορά που χτίζεται ακόμα και ένα σχολείο, να προβλέπεται η διευκόλυνση των ατόμων με αναπηρία. Οφείλει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση να συνάδει πλέον με την Σύμβαση Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Τόπων με Αναπηρίε και η αξιολόγηση τη σύμβαση αυτή πλέον και τη συμμόρφωση Ευρωπαϊκή Ένωση γίνεται μέσω τη γνωμοδότηση που θα εξετάσουμε σε λίγο. Θα ήθελα να περάσω τώρα στο κείμενο τη γνωμοδότηση αυτή. Θεωρώ ότι η πρωτοβουλία αυτή καταρχά είναι αξιέπαινη πολύ σημαντικό το ότι αποφασίσετε εσείς να υποβάλλετε προς την Επιτροπή Απασχόλησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μια τέτοια γνωμοδότηση. Θεωρώ ότι μέσω της γνωμοδότησης αυτής μπορείτε εσείς ως Επιτροπή Ανάπτυξης να ενισχύσετε την εξωτερική πτυχή αυτής της πολιτικής, να υπενθυμίσετε τελικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι η προώθηση των δικαιωμάτων των ατόμων αναπηρία δεν έχει να κάνει μόνο με τις εσωτερικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά θα πρέπει να υφίσταται και να προωθείται και σε όλες τις εξωτερικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η δική σας η Επιτροπή φέρει την αρμοδιότητα αυτή. Θα ήθελα να κάνω τρεις συγκεκριμένε προτάσεις όσον αφορά το κείμενο τώρα της γνωμοδότησης. Καταρχάς, θα πρέπει θεωρώ να συμπεριλάβετε μια σύντομη αναφορά στο πλαίσιο πολιτικής ε, που ε, ακολουθείται με ορίζοντα το 2030, ιδίω όσον αφορά την ανθρωπιστική βοήθεια και όσον αφορά τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης. Νομίζω λοιπόν ότι θα ευθυγραμμιστεί καλύτερα το κείμενο αν κάνετε μια τέτοια μνήμα. Δεύτερη παρατήρηση, δεύτερη προσθήκη που θα πρότεινα, να αναφέρεται επίση το ρόλο που δραματίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση κατά την προώθηση τη σύμβαση αυτή των Εθνών, ιδίω μέσω διαφόρων μορφών διαλόγων που έχει με διάφορε χώρε. Αναφέρομαι σε διάλογο που μπορεί να έχει να κάνει με τα ανθρώπινα δικαιώματα, με την ανθρωπιστική βοήθεια ή διάλογο που μπορεί να έχει να κάνει με την αναπτυξιακή βοήθεια και να αναφερθείτε επίσης και στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθώντας να εφαρμόσει τη σύμβαση αυτή. Σε καμία περίπτωση αυτή τη στιγμή δεν θέλω να δώσω την εντύπωση ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αντιμετωπίζει κανένα πρόβλημα. Είναι πολύ σημαντικό να αντιμετωπίζουμε και τα προβλήματα τα οποία προκύπτουν κατά τη διάρκεια των διεθνών αυτών διαλόγων. Και να βλέπουμε επίσης πώς συμβάλλουν και οι χώρες αποδέκτες στα πλαίσια του διαλόγου αυτού. Τρίτη και τελευταία τώρα παρατήρηση που θα ήθελα να κάνω πάντα προς το κείμενο της γνωμοδότησης είναι ενδεχομένω να κάνετε μία αναφορά στις ε, υφιστάμενες ή μελλοντικέ ε, δυνατότητες πολιτικής που θα έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση στον τομέα αυτό. Να φερθώ σε δύο συγκεκριμένες. Πρώτον, το η νέα επαναδιατυπωμένη, αναθεωρημένη συνένεση για την ανάπτυξη. Ξέρετε ότι αυτό είναι ένα από τα βασικότερα υψηλόβαθμα κείμενα, τα οποία διασφαλίζουν ότι όντως μπορούμε να έχουμε ευθυγράμμιση των πολιτικών μας και ότι θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και η διάσταση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να γίνεται μία αναφορά και σε αυτό το κείμενο της ε, συνένεσης αυτής και επίσης να γίνεται και μία αναφορά στην ε, ενδιάμεση αναθεώρηση του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου, καθότι θα μπορούσαμε να δούμε από χρηματοοικονομικής, ε, δημοσιονομικής πλευράς τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν δεσμεύσεις όσον αφορά την ένταξη της διάταξης των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία στον απτυξιακό τομέα. Ας δούμε λοιπόν από οικονομικής πλευράς τι όντως έχει κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση και τι κονδύλια προβλέπεται να δεσμεύσει στο μέλλον. Ολοκληρώνοντας κάτι ακόμα να σας πω. Θεωρώ ότι ουδέποτε μέχρι σήμερα δεν είχαμε ένα τόσο ισχυρό πάγιο πλαίσιο για την ε, υλοποίηση, την πραγμάτωση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία. Αναφέρθηκα σε διάφορες συμφωνίες, σε διάφορα πλαίσια που είχαμε στο παρελθόν. Αυτή τη στιγμή όμως έχουμε ένα πολύ ισχυρό κείμενο το οποίο πρέπει να εφαρμοστεί. Οι δεσμεύσει θα πρέπει να γίνουν πραγματικότητα. Συμμετέχει προφανώς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, συμμετέχουν οργανώσεις που εκπροσωπούν την κοινωνία των πολιτών όπως η δική μου, ρόλος μας θεωρώ είναι να παρακολουθούμε την εφαρμογή των δεσμεύσεων αυτών και να επενθυμίσουμε στους υπεύθυνου χάραξης πολιτικής ότι ε, η απλή αναφορά των ατόμων με αναπηρία σε διάφορες συμφωνίες δεν ε, διασφαλίζει το ότι όντω προασπίζονται τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία. Ανταυτού θα πρέπει να ασκούμε συνεχή πίεση προκειμένου να προασπίζονται τα δικαιώματα αυτά. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Εγώ και εγώ σας ευχαριστώ. Πρώτα η κυρία Χάουταλα που είναι και η συγγήτρια της εκθέσεως. Ευχαριστώ Λίντα. Όσα είπε ο κύριος Μπόσελμαν είναι απολύτως ορθά. Και συμφωνώ απόλυτα στην ανάγκη να περιληφθεί η ε, να περιληφθούν δηλαδή οι ανάγκες των ανθρώπων με ειδικέ ανάγκες σε, όλες, σε όλους τους πολιτικής. Είχαμε και ειδική συνεδρία για την αναπηρία και ακούσαμε πολλούς εκπροσώπους κυβερνήσεων μετέφεραν το μήνυμα των αναπήρων που λένε μην αποφασίζετε τίποτα χωρίς τη δική μας συμμετοχή. Οι άνθρωποι παίζουν ρόλο και στη διαμόρφωση των πολιτικών για να είναι η ζωή τους ίση με την ζωή των υπολείπων. Επίσης, εξ όσων είπε ο κ. Μπόσελμαν, για την Σύμβαση για τα Δικαιώματα Ανθρώπων με Αναπηρίες, είναι μια πραγματικά μοναδική ευκαιρία για να επιφέρουμε τις αλλαγές από, όπως είπα, τους και ούτω Προ όχι πολλού χρόνου έπεσα σε μια ιστοσελίδα των Ουκρανικών Διεθνών Αερογραμμών που έλεγαν ότι ανάπηροι άνθρωποι έχουν πρόσβαση στις πτήσεις τους αλλά εάν κάτι από την παρουσία τους ενοχλεί τους υπόλοιπους επιβάτες μπορούν να τους διώξουν από την πτήση. Είναι δυνατόν. Πώς ε, ε μπορεί να επαναληφθεί κάτι τέτοιο. Πολύ ευχαρίστω να συνεργαστώ με τον κύριο Πόσελμαν που εκπροσωπεί μια μεγάλη, ένα μεγάλο συνασπισμό ανθρώπων που ε, έχουν απειρίες και τις οργανώσεις τους για να βελτιώσουμε τη γνωμοδότηση και να διασφαλίσουμε ώστε η αναπηρία με όλες τις διαστάσεις της να ενταχθεί πλήρως σε όλους τους τομείς πολιτικής της Ένωσης καθώς και ε, αναπτυξιακής πολιτικής κλπ. Μπορούν να γίνουν πολλά πράγματα. Χαίρομαι που αναφέρθηκε και το Σέντα πλαίσιο για την αντιμετώπιση καταστροφών και ε, αυτό θα πρέπει να το προσθέσουμε επίσης. Δεν νομίζω ότι έχω να προσθέσω τίποτε περισσότερο. Πρέπει να διασφαλίσουμε ώστε η Επιτροπή Αναπτύξεως να τονίσει ιδιαίτερα την διάσταση αυτή της αναπτυξιακής πολιτικής και όπως είπε ο κ. Μπόσελμαν να επιμείνουμε ώστε η αναπηρία να αποτελέσει ε, θέμα σε όλους τους διαλόγους μεταξύ Ευρωπαϊκής Ενώσεως και των εταίρων της. Και ένας από τους καλύτερους τρόπους για να βελτιώσουμε τη ζωή των ε, αναπήρων στις αναπτυσσόμενες χώρες είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση να δώσει περισσότερη στοχευμένη ενίσχυση για τις κινήσεις των ίδιων των αναπήρων. Μάλιστα. Νταβό Στίερ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εσάς κύριε πόσελμαν. Εγώ θα ήθελα ωστόσο να συνεχίσω, να αφήσω τα αγγλικά δηλαδή και να συνεχίσω τα κροατικά, οπότε φορέστε τα ακουστικά σας. Έλεγα λοιπόν ότι ευχαριστώ τον κύριο Μπόσελμαν για τα σχόλιά του και τις προτάσεις του για την, ε, σχετικά δηλαδή με τη γνωμοδότηση την οποία θα συντάξουμε και θα ψηφίσουμε στην Επιτροπή μας. Πιστεύω όντως ότι θα εκπροσωπήσουμε τα ενδιαφέροντά σας αυτά εδώ. Πρώτα έχω ένα γενικό σχόλιο για τους νομικούς ορισμούς που έχουν άμεσες επιπτώσεις. Γνωρίζω για τα προβλήματα των κοφαλάλων που είναι προβλήματα τα οποία καμιά φορά ούτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι αρκετά ξεκάθαρα ορισμένα από νομική σκοπιά. Σε ορισμένες χώρες δεν διαθέτουν δικαιώματα ή τέλο πάντων δεν μπορούν να απολαύσουν ε, τα δικαιώματά τους οι κοφάλαλοι διότι δεν υπάρχουν σχετικέ οργανώσει κλπ. Το ίδιο ισχύει και για χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεύτερη παρατήρηση. Αναφερθήκατε στο ότι θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε την ευκαιρία που μας ανοίγει αυτή η δημιουργία συνένεσης για την ανάπτυξη. Δικέ μου πληροφορίε που λένε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προβεί σε δημοσίευση ανακοινώσεως περί τα τέλη του έτου. Χθες έλαβα πιο ενημερωμένε πληροφορίε, που λένε όμως ότι μάλλον περιμένουμε μέχρι τι αρχέ του 2017. Αυτό ίσως είναι ενδιαφέρουσα πληροφορία για σας και για την κοινωνία των πολιτών γενικότερα. Οι πληροφορίε δηλαδή αυτέ που έχω λένε ότι την επόμενη εβδομάδα θα αρχίσει η δημόσια διαβούλευση για την εσωτερική και εξωτερική εφαρμογή των νέων παγκόσμιων στόχων της Ατζέντα 2030. Και κάποια στιγμή τον Νοέμβριο του 2016 θα εκδοθούν δύο ανακοινώσεις. Μία για τις εσωτερικές ε, εφαρμογές της ε, ε, ατζέντα των αναπτυξιακών στόχων και εντός, και εντός, εκτός της Ένωσης και θα είναι σημαντικό να ακουστούν και οι απόψεις της κοινωνίας των πολιτών και των οργανώσεων σας. Και μετά από αυτό το 2017 πλέον θα εκδοθεί σχετική ανακοίνωση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για αυτή τη νέα αναπτυξιακή συνένεση. Αυτές τις προφορές έλαβα εχθέ και ελπίζω ότι είναι χρήσιμες για σας. Ευχαριστώ. Σλάιν. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Μιλώ τώρα εξ ονόματος συναδέλφου Πατρίτσια Τόια. Ε, ακούμε ένα θόρυβο από το μικρόφωνο σας. Υπάρχει κάποια παρέμβαση. εντάξει, διορθώθηκε. Έχετε το λόγο. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω τη συνάδελφο αλλά εξ ονόματος τη συναδέλφου Πατρίτσια Τόια, η οποία δεν μπορεί να παρευρίσκεται εδώ πέρα σήμερα και μου ζήτησε να διαβάσω ένα σύντομο σημείωμα. Σεστό λοιπόν συγγνώμη που δεν μπορώ να έρθω σήμερα, αλλά έπρεπε να επιστρέψω στην Ιταλία για μια σημαντική συνάντηση που έχω στην πόλη μου το Μιλάνο. Θεωρώ όμω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό η Επιτροπή Ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να καταφέρει να γνωμοδοτήσει όσον αφορά την εφαρμογή της Σύμβασης Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες. Θα πρέπει να θυμάμαστε ότι ένα 15% του παγκόσμιου πληθυσμού, περίπου δηλαδή ένα δισεκατομμύριο άτομα, ζουν με μια κάποια αναπηρία και περίπου το 80% των ανθρώπων αυτών βρίσκονται σε φτωχές συναπτυσσόμενες χώρες. Πρέπει λοιπόν αυτό να το έχουμε κατά νου. Στις τροπολογίες που πρόκειται να καταθέσω θέλησα να τονίσω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξεκινήσουν συγκεκριμένε δράσεις mainstreaming, ζήτημα το οποίο είναι θεμελιώδου σημασίας προκειμένου να καταφέρουμε να έχουμε μια βιώσιμη ανάπτυξη που θα περιλαμβάνει τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία. Θα πρέπει να έχουμε τους απαραίτητους μηχανισμούς για τη συλλογή και την παρακολούθηση μη ενοποιημένων δεδομένων όσον αφορά την ηλικία, την αναπηρία συγκεκριμένων ατόμων που υπάγονται σε πολιτικές αναπτυξιακής συνεργασίας. Η έλλειψη στατιστικών δεδομένων αυτή τη στιγμή καθιστά τη δική μας τη δράση μη αποτελεσματική, ιδίω όσον αφορά την πρόθεση των δικαιωμάτων ατόμων με αναπηρία στις αναπτυσσόμενες χώρες. Είναι πολύ σημαντικό να καταφέρουμε να υποστηρίξουμε τα άτομα όχι μόνο σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, αλλά κυρίως την περίοδο μετά από, την, μετά από μια καταστροφή, μετά από μια επίγουσα κατάσταση. Ευχαριστούμε πολύ. Θέλετε να απαντήσετε σε όλες αυτές τις ερωτήσεις. Σας ευχαριστώ πολύ. Ακούσαμε ερωτήσεις, αλλά ακούσαμε και κάποιες γενικές παρατηρήσεις. Όσον αφορά τον δικό μου τον οργανισμό και ξεκινώντας με την τελευταία παρατήρηση, συμφωνώ και εγώ ότι δεν πρέπει να έχουμε μόνο ομαδοποιημένα, ενοποιημένα δεδομένα, αλλά θα πρέπει να έχουμε και πιο λεπτομερή επιμέρους δεδομένα όσον αφορά τις συγκεκριμένε αναπηρίες. Αυτό το βλέπουμε και στην Ατζέντα 2030. Εκφράζεται μια τέτοια απέτηση. Αυτό όμως προϋποθέτει μια πολύ σημαντική διοικητική ικανότητα όσον αφορά τις στατιστικές αρχές των ε, χωρών και ιδίω των φτωχών χωρών. Μας έχει απασχολήσει πάντως το ζήτημα αυτό και έχετε απόλυτο δίκιο που το θίγετε, γιατί τα ποσοστά στα οποία αναφερθήκατε 15% και στη συνέχεια το 80% αυτού του 15% αντιστοιχούν σε πολύ μεγάλο αριθμό ανθρώπων για τους οποίους δυστυχώς έχουμε μόνο κάποιες εκτιμήσεις. Ακόμα και τα ποσοστά αυτά δεν είναι εντελώς αξιόπιστα στατιστικά δεδομένα, αλλά κάποιες αρχικές εκτιμήσεις. Όσον αφορά τώρα τη συνένεση για την ανάπτυξη. Σας ευχαριστώ για τη σχετική σας παρατήρηση και για τις πληροφορίες που μας δώσατε. Δεν γνώριζα αυτά τα οποία είπατε, ότι θα πρέπει δηλαδή να συνεχιστούν οι προσπάθειες και του χρόνου, ότι δεν πρόκειται δηλαδή το σχετικό εγχείρημα να ολοκληρωθεί φέτος. Αν δεν κάνω λάθος, όμως ήδη το Μάιο προβλέπεται σε υπουργικό επίπεδο μία συζήτηση μεταξύ των Υπουργών Ανάπτυξης. Να μία περαιτέρω πληροφορία που μπορώ να σας δώσω και ελπίζω ότι είναι σωστή. Πάντως, σας διαβεβαιώ ότι εμείς θα παρακολουθούμε εκ του σύνεγγυ στην όλη διαδικασία και θα προσπαθήσουμε να συμβάλλουμε και σε όλες τις μορφές διαβούλευσης που θα λάβουν χώρα προκειμένου να καταλήξουμε στο οριστικό αυτό κείμενο για τη συνένεση για την ανάπτυξη. Όχι μόνο επειδή είναι σημαντικό να υπάρχει ως κείμενο, αλλά επειδή τελικά θα είναι ένα έγγραφο το οποίο θα παρουσιάζει όλες τις διαφορετικές απόψεις όλων των διαφορετικών φορέων και κυβερνήσεων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα αυτό αναπτυξιακής συνεργασίας ολοκλήρωσε τις παρατηρήσεις μου σε αυτό το σημείο. Σας ευχαριστούμε πολύ. Για πρώτη φορά βλέπουμε ίσως να κάνει περισσότερα πράγματα το Συμβούλιο από ότι εμείς θέλαμε να ενημερωθούμε για το τι γίνεται σε επίπεδο Συμβουλίου. Η Παθιένθια η Μακουλάδα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, παρακαλώ. Αλλά όχι για πολλή ώρα, παρακαλώ. Ναι, θα είμαι πολύ σύντομη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για την υλοποίηση της ε, Σύμβασης των ΗΠΑ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία και χαιρετίζει τη σημερινή συζήτηση καθώς και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής σας στην έκθεση της Επιτροπής Απασχόλησης. Θα ήθελα να υπογραμμίσω ε, ότι η πρόθεση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία στο πλαίσιο των εξωτερικών δράσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι και ένας από τους στόχους της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τα άτομα με αναπηρία για το 2014-2020 περιλαμβάνει τις εξωτερικές δράσεις ε, και αυτή τη φάση ε, κάνουμε έναν απολογισμό και προετοιμάζουμε την έκθεση πεπραγμένων σε σχέση με τη στρατηγική αυτή και θα συμπεριλάβουμε στοιχεία που θα αφορούν τις δραστηριότητες που οποίο αναφέρονται σε αυτή τη στρατηγική καθώς και θα εξετάσουμε τα συμπεράσματα, τις καταληκτικές παρατηρήσεις της Επιτροπής EPRD μετά το διάλογο με την Ευρωπαϊκή για την εφαρμογή της σύμβασης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Θέλει να πει κάτι η Χάιντι. Ναι, πολύ σύντομα. Να πω ότι πιστεύω ότι έχουμε πολλά, ε, δυνατότητες με τις τροπολογίες μας να βελτιώσουμε την έκθεση αυτή και τις Περιμένω με ενδιαφέρον, φέσα και από την κοινωνία των πολιτών, τον κύριο Πόστονα και άλλους, 25 Απριλίου, την ε, Δευτέρα δηλαδή που μα έχετε ε, λίγη προθεσμία στο 12 το μεσημέρι, άρα γρήγορα να κάνετε παρακαλώ. Ναι, αυτό θα έλεγα λέει πρόεδρο. 25 Απριλίου είναι η καταληκτική προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών. Θα ψηφίσουμε στις 24 Μαΐου. Να ευχαριστήσω τον κύριο Μπόσελμα που ήρθε εδώ και μας διαφώτισε και ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να κάνουμε ένα βήμα προς σωστή κατεύθυνση για να εξασφαλίσουμε αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης για όλα τα άτομα με αναπηρία. And I'll invite um, Eric εσείς ελάτε τώρα εδώ. Okay, Φτάνουμε στο υπαριθμό 20 για την μέτρηση ODA. Έχουμε κοντά μας τον Έριχ Σόλχαϊμ, πρόεδρο της Επιτροπής Αναπτυξιακής Βοήθειας του ΟΣΑ. Έγινε ήδη συνεδρία της Επιτροπής αυτής τον Φεβρουάριο στο Παρίσι. Έχουν ληφθεί αποφάσεις για την αλλαγή του τρόπου με τον οποίο λειτουργεί. Γνωρίζετε σίγουρα, Έρικ, ότι πολλοί θέτουν υπόψη μας τις ανησυχίες, τις ανησυχίες τους για τις αλλαγές στο ODA που θα ε, ε, επιτρέπουν το άνοιγμα του reporting του ODA για τη χρηματοδότηση στρατιωτικού προσωπικού το οποίο ε, αποδυναμώνει τα όρια μεταξύ αναπτυξιακής βοήθειας και χρηματοδοτικής ενίσχυσης στρατιωτικών δυνάμεων. Κατανοούμε βέβαια το θέμα, αλλά ποιος είναι ο προβληματισμός. Προφανώς υπάρχει πίεση και λόγω μεταναστευτικής κρίσης επί της ODA και επειδή και πολλές ε, χώρες, πολλές κυβερνήσεις δηλαδή δαπανούν χρήματα για το μεταναστευτικό και μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι γίνεται με αυτό. όπου ODA σημαίνει επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια. Ε, έτσι λοιπόν ε, συζητήσαμε κιόλας και μεταξύ μας και με την ε, Νότια Αφρική και μιλήσαμε και για τη συνεργασία, για τα έγγραφα Παναμά και την αναπτυξιακή βοήθεια κτλ. που είναι όλο και περισσότερο γνωστά και είναι χρήσιμη η ε, παρουσία σας σήμερα εδώ για να μας εξηγήσετε τα σχετικά. Σας ευχαριστώ πολύ αγαπητή Λίντα. Με χαρά επανέρχομαι ενώπιόν σας της Επιτροπής Αναπτύξεως της Ευρωβουλής να σας εξηγήσω πρώτα την ευρύτερη εικόνα και να συζητήσουμε τις λεπτομέρειες μετά. Η ευρύτερη εικόνα έχει ως εξής. Το μέγα μυστικό που είναι και καλά κρυμμένο εδώ στην Ευρώπη, ο κόσμος είναι ένας πραγματικά θαυμάσιος κόσμος, αγγελικά πλασμένος και ε, βρισκόμαστε σε μια από τις ευτυχέστερες στιγμές της ανθρώπινης ιστορίας. Το 2015 ήταν το τυχερότερο έτος στην ανθρώπινη ιστορία για το απλό άνθρωπο. Βεβαίω ε, δεν θα συμφωνήσουν όλοι στην Συρία για παράδειγμα, αλλά για τον μέσο άνθρωπο η κατάσταση στον πλανήτη ποτέ δεν ήταν καλύτερη από ε, την χρονική αυτή περίοδο που διανύουμε. Οι άνθρωποι ε, είναι πιο μεγαλόσωμοι, καλύτερα, ε, διατρέφονται καλύτερα, έχουν καλύτερη εκπαίδευση, καλύτερη υγεία και ούτω καθεξής. Το 2015, πέρσι δηλαδή, ήταν αυτό που σας είπα, το 2016, Αυτά. Νούμερα. 7 εκατομμύρια. Ένας αριθμός που μπορείτε να θυμάστε. Ο αριθμός των παιδιών που επέζησαν το 2015 γιατί έχουμε μειώσει την παιδική θνησιμότητα, την έχουμε μειώσει στο μισό. Και αυτό καθιστά πολλούς γονείς ευτυχισμένους. Φανταστείτε, αυτά τα παιδιά θα είχαν χάσει τη ζωή θα είχαν Βέβαια αυτά μπορεί να μην είχαν απασχολήσει όλα τα διεθνή μέσα ενημέρωση, αλλά θα ήταν ένα μέγα δράμα για του γονεί του. Τώρα, υπάρχουν δύο λόγοι για τους οποίους θα πάμε καλύτερα. Πάλι η ευρύτερη εικόνα από τον Αδάμ και την Εύα μέχρι το 1990 είχαμε κάθε χρόνο περισσότερους ανθρώπους στον πλανήτη. Από την απαρχή της βιομηχανικής επανάστασης στο Μάντσεστερ και μέχρι το 1000 Άρχισε να μειώνεται όμως μετά ο ο αριθμό, η αύξηση, ο ρυθμός της αύξησης δηλαδή, έχουμε μειώσει τις ασθένειες, έχουμε μειώσει θανάτου από ασθένειες, την παιδική θνησιμότητα κλπ. Υπάρχουν δύο λόγοι. Καλύτερες πολιτικές, περισσότεροι πόροι. Οι πολιτικές είναι και πιο σημαντικές. Οι μεγάλες επιτυχίες των, ε, του Σιγκαπούρης και ούτω καθεξής είναι διότι έχουν εφαρμόσει ορθές πολιτικές. Όχι επειδή έχουν περισσότερους πόρους, εξετάστε και την Αφρικανική Ήπειρο, θα δείτε αύξηση της τάξης των 10% τον χρόνο τα τελευταία 15 χρόνια. Άρα, η εφαρμογή ορθών πολιτικών είναι το νούμερο ένα και χρειαζόμαστε ένα συνδυασμό ισχυρών κρατών, να αποφύγουμε δηλαδή το, την λάθος σκέψη των ακροδεξιών ότι μπορούμε να καταργήσουμε το κράτος και να αποφύγουμε και το ε, ε λάθος της ακροαριστεράς σκέψης που, που λέει ότι μπορούμε να ξεφορτωθούμε τις αγορές και θα τα καταφέρουμε μια χαρά. Και τα δύο αυτά είναι λάθος. Και το άλλο είναι η πόρη. Στην Αντισαμπέμπα πέρσι είδαμε ότι υπάρχουν τρεις βασικοί πόροι. Φόροι, ιδιωτικές επενδύσεις και αναπτυξιακή βοήθεια. Από αυτά τα τρία, οι φόροι είναι οι πιο σημαντική. Εμεί θεωρούμε εδώ στην Ευρώπη ότι η ανάπτυξη προέρχεται από τι δικέ μα προσπάθειε. Α, η εκπαίδευση λένε ορισμένοι που προσφέρει η UNICEF, η Ευρωπαϊκή Ένωση ή δεν ξέρω ποιο άλλο. Όχι, ξεχάστε τα αυτά. 98 και παραπάνω τη 100 από την εκπαίδευση τη αναπτυσσόμενη χώρα πληρώνεται από του φορολογούμενου των χωρών αυτών. Οι φορολογούμενοι τη Κίνα πληρώνουν για την παιδεία στην Κίνα. Στην Ινδία το ίδιο, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η διεθνής κοινότητα δεν παίζει σημαντικό ρόλο. Προσφέρουμε τεχνολογία, τεχνογνωσία, βέλτιστες πρακτικές και άλλα αγαθά. Όμως, το βασικό βάρος το σηκώνουν στους ώμους τους οι φορολογούμενοι των χωρών αυτών. Επομένως, οι φόροι παίζουν σημαντικό ρόλο. Γι' αυτό ήρθε εδώ και ο Ταμπομπέκη. Τα χρήματα φεύγουν από την Αφρική, τα είδαμε αυτά, σε δεκαπλάσιο ρυθμό από αυτά που πηγαίνουν στην Αφρική. Αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί. Είναι τεράστια η ζημιά για τους λαούς των χωρών της Αφρικής. Και είναι όμως και ανέντιμο απέναντι στους άλλους φορολογούμενους. Γιατί να προσφέρουν τα χρήματά τους για να αναπτυξιακή βοήθεια στην Αφρική όταν αυτά και πολύ περισσότερα εξέρχονται πάλι της Αφρικής για να φτάσουν σε φορολογικούς παραδόσεις. Αυτό πρέπει να σταματήσει λοιπόν. Γι' αυτό έχουμε ξεκινήσει τώρα ένα μεγάλο αριθμό ε, πρωτοβουλειών για να βελτιώσουμε τα φορολογικά συστήματα. Εστιάζουμε τώρα σε τούτην εδώ την πρωτοβουλία που ενισχύει τις χώρες για να στήσουν αποδοτικά φορολογικά συστήματα. Το έστω το 10% ενώ στην Ευρώπη είναι 35%. Η διαφορά είναι μεγάλη. Χρειαζόμαστε λοιπόν καλύτερε φορολογικέ διοικησει στις αναπτυσσόμενες χώρες. Τα επόμενα χρόνια θα έχουμε και αυτόματε ανταλλαγέ φορολογικών στοιχείων. Άρα η νορβηγική κυβέρνηση τη Πατρίδα μου δηλαδή μπορεί να ρωτήσει την, ε, τις φορολογικές διοικήσεις του ε, Ηνωμένου Βασιλείου ή τη Ελβετία ή του Λουξεμβούργου, δεν ξέρω πού αλλού, για να λάβει τα στοιχεία που τις χρειάζονται για τις έρευνε τη. Θα είναι πιο δύσκολο για τις χώρες εκείνες που δεν έχουν πραγματική ε, αποδοτική φορολογική διοίκηση να χρησιμοποιήσουν πληροφορίες αυτές. Γι' αυτό και πρέπει να ενισχυθεί η συνεργασία. Και η αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών και δεδομένων και μετακινήσεων κεφαλαίων δηλαδή θα ενισχύσει πολύ. Τώρα έχουμε και αυτό το BEPS που σημαίνει ε, ε, διάβρωση της φορολογικής βάσης και μεταφορά κερδών. Δεν είναι καταρχήν παράνομο, όπως είπε όμως ο Μπαράκ Ομπάμα δεν ενδιαφέρει είναι παράνομο, είναι σαφώς ανήθικο. Μετακινείτε λοιπόν τα κέρδη σας κάπου όπου δεν χρειάζεται να πληρώσετε φόρους αντί να φορολογηθείτε εκεί όπου είναι η παραγωγή, σα. σας. Ο δε Υπουργός Οικονομικών Όσμπορν της ε, Μεγάλης Βρετανίας επιτέθηκε κατά Starbucks, Google και ε, Apple που δεν πληρώνουν φόρους στο Ενωμένο Βασίλειο. Δεν πληρώνουν φόρους ούτε στο Βιετνάμ ούτε στο Περού πάνε και εγκαθίστανται στον Παναμά. Χρειάζεται λοιπόν να ανακόψουμε την πορεία αυτή. Οι φόροι θα πρέπει να καταβάλλονται εκεί όπου είναι η παραγωγή του προϊόντος. Εάν έχετε πλοίων τόπους όπου παράγεται το προϊόν, θα πρέπει να πληρώσετε και στο Κονγκό και στο Βέλγιο και δεν ξέρω που αλλού. Υπάρχουν και άλλες πολλές πρωτοβουλίες. Εσείς ως πολιτικοί άνδρες και γυναίκες έχετε και το μεγαλύτερο δώρο στην ανθρώπινη ιστορία. Έχετε την ευκαιρία να χρησιμοποιήσετε τις δυνατότητες αυτές για να μειωθούν ε, η φορολογική παράδοση, η παράδοση, να ε, καταργηθούν. Πρόκειται για μια τεράστια ευκαιρία και δεν πρέπει να χάσετε την ευκαιρία να βάλετε τον κόλ. δεν πρόκειται μόνο για θέμα πολιτικής βούλησης στην Ευρώπη, στις ΗΠΑ, της Αμερικής, στην Κίνα, στις άλλες μεγάλες χώρες του κόσμου. Πρέπει να εκμεταλλευτείτε την ευκαιρία. Πρέπει να εκμεταλλευτούν οι πολιτικοί την ευκαιρία. Χαμηλό επίπεδο φορολογίας, αλλά κάποιοι πρέπει να πληρώνουν για να φύγει ο κόσμος από την φτώχεια. Και η φόροι, επαναλαμβάνω, είναι ο βασικός συντελεστής της ανάπτυξης. Δεύτερο, βεβαίως, οι ιδιωτικές επενδύσεις. δηλαδή ε, για την επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια. Πώς μπορούμε να την εκμεταλλευτούμε καλύτερα. Αν θέλετε να υλοποιήσετε τα υπεσχημένα της Συμφωνίας των Παρισίων, πρέπει όλες οι χώρες να συνεργαστούν. Μια πάρα πολύ μεγάλη, μια πάρα πολύ σημαντική συμφωνία στην ανθρώπινη ιστορία. Αν θέλουμε να τηρήσουμε τα υπεσχημένα λοιπόν, είναι πολύ σημαντικό να γίνουν επενδύσεις στο πράσινο κοινοτήμα της οικονομίας. Τώρα για την επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια που είναι αυτό που μπορεί να αλλάξει τις ροές. Για τις πιο φτωχές χώρες του πλανήτη είναι πολύ σημαντική, διότι πρόκειται για τα δύο τρίτα των εισρώων στις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες. Είναι ακόμα περιορισμένα όμως ε, τα ποσά αυτά για χώρες όπως Βραζιλία, ε, Ινδίες, ε, Τουρκία κλπ. Χρειάζεται λοιπόν να στοχεύσουμε την αναπτυξιακή βοήθεια περισσότερο προς τις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες και λιγότερο προς τις χώρες μέσου εισοδήματος. Κάνουμε βήματα για την επίτευξη του στόχου αυτού. Το 2015 για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια ε, έσπασε αυτή η ε, τάση, η πτωτική τάση των ε, επενδύσεων προς τις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες και άρχισε να αυξάνεται και πάλι. Δεν έχει μειωθεί η αναπτυξιακή βοήθεια ούτε στη διάρκεια της δημοσιονομικής κρίσης, ούτε στη διάρκεια της ανθρωπιστικής κρίσης και τώρα που το μεταναστευτικό έχει μπει και το προσφυγικό έχει μπει στην κορυφή τη πολιτική ατζέντα αυξάνεται διαρκώς τα τελευταία χρόνια η αναπτυξιακή βοήθεια. Όμω δεν φτάνει στα επίπεδα που έχουν υποσχεθεί οι χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλε χώρε ανά τον κόσμο. Δεν έχει φτάσει στο επίπεδο αυτό, όμως αυξάνεται κάθε χρόνο και πρέπει να προσανατολιστεί, να κατευθυνθεί περισσότερο προς τις λιγότερο αναπτυγμένε χώρε. και να χρησιμοποιηθεί περισσότερο ω καταλήτη για άλλου θετικού σκοπού. Αυτά είναι τα πράγματα που αναφέρατε και εσεί προηγουμένω. Υπάρχουν τέσσερις μείζονες μεταρρυθμίσεις που προσπαθήσαμε να επιφέρουμε τα τελευταία χρόνια σε ό,τι αφορά την χρήση της ε, επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας, όπως είπα, με κατεύθυνση περισσότερο από τις, προς τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες. Βεβαίως, η ιδιωτική επένδυση δεν πρόκειται να προσφέρει παιδεία. Αυτά είναι φαντασίες. Υπάρχουν κάποια πράγματα που μπορεί να λάβει μόνο ο δημόσιος τομέας. Η μικρότερη και λιγότερο σημαντική αλλαγή είναι η αλλαγή κάποιων κανόνων σχετικά με την ειρήνη και την ασφάλεια. Πολύ μικρές αλλαγές που ίσως αφορούν το 1% της βοήθειας. Πολύ μικρή σημασία για το συνολικό όγκο της αναπτυξιακής βοήθειας. Όμως κάποιες οργανώσεις Τη ε, κοινωνία των πολιτών φοβούνται ότι περισσότερη αναπτυξιακή βοήθεια θα κινηθεί προς τη χρηματοδότηση στρατιωτικών δυνάμεων. Αυτό είναι λάθος. Εγώ ήμουν και 7 χρόνια στο Νορβηγικό Αρμόδιο Υπουργείο και αν υπήρχε έστω... Δεν υπάρχει ούτε μία πιθανότητα, τέλος πάντων, ο ε, Υπουργό Ανάπτυξη στην Νορβηγία να δεχθεί να πάνε κάποια κονδύλια σε στρατιωτικέ δυνάμει, για παράδειγμα το Αφγανιστάν. μπορεί η σκοπή αυτή να είναι χρήσιμη διότι η ασφάλεια ε, παίζει ρόλο κλειδί για την ανάπτυξη, από την άλλη μεριά όμως θα υπονομεύσει για παράδειγμα την υγεία και την παιδεία. Απάντησε η ανταπόκριση του Ηνωμένου Βασιλείου στην κρίση του ιού έμπολα ήταν πολύ σημαντική. Στήριξε τους ε, ιατρούς χωρίς σύνορα και άλλες οργανώσεις. Πάρα πολύ σημαντική η προσπάθεια αυτή. Το Ηνωμένο Βασίλειο θέλησε να στείλει στρατιωτικά νοσοκομεία στην περιοχή αυτή και αυτό έγινε χωρίς πρόβλημα. Και χρησιμοποίησε γι' αυτό πανάκριβες εταιρείες charter. Θα μπορούσε να έχει χρησιμοποιήσει στρατιωτικά αεροσκάφη πολύ φθηνότερα και πολύ ταχύτερα. Αυτό δεν θα ήταν, ωστόσο, δεν θα αναγνωριζόταν ως βοήθεια. Εμείς το βρήκαμε παράλογο αυτό και θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί στο μέλλον καλύτερα. Από την άλλη μεριά είναι ευκολότερο να εκπαιδευτεί το στρατιωτικό προσωπικό για την αντιμετώπιση βίας κατά προσώπων στην βάση του φύλου και ούτω καθεξής. Αλλά όπως είπα πρόκειται για πολύ μικρές αλλαγές. Δεύτερη αλλαγή που κάναμε νομίζω ότι τα έχουμε ξαναπεί στην Επιτροπή σας, για τα δάνεια. Οι ευρωπαϊκές χώρες προσφέρουν χρήσιμα δάνεια για την ανάπτυξη. Αλλάξαμε τους κανόνες τώρα, ώστε ένα δάνειο που προσφέρεται σε μια ελάχιστα ανεπτυγμένη χώρα να μετρά περισσότερο από ένα δόνιο, δάνειο συγγνώμη, το οποίο ε, προσφέρεται σε μια χώρα μέσου εισοδήματος. Αλλάξαμε τους κανόνες λοιπόν, ώστε να έχετε αυτό το ισοδύναμο επιχορήγησης, grand equivalent δηλαδή, που μπορεί να θεωρηθεί κρατική ενίσχυση, διότι στο παρελθόν το σύστημα ήταν ότι αν η συμπεριφορά σας δεν ήταν σωστή για ένα θάνιο δεν, ε, πιστονός, ε, δεν λαμβάνατε καμιά πίστοση γι' αυτό. Και τέλος πάντων ε, ε, ε, τα κίνητρα ήταν λάθος στην περίπτωση αυτή. Τρίτο, ε, ρίξαμε ιδιαίτερα την προσοχή μας στον ιδιωτικό τομέα. Διάφορες χώρες μέλη της Ένωσης έχουν διαφορετικά συστήματα και το σύστημα που εφαρμόζουμε τώρα είναι ότι οι χώρες αυτές όπως το Ηνωμένο Βασίλειο και οι σκανδιναβικές χώρες έχουν αναπτύξει δημοσιονομικούς θεσμούς και αυτοί η βοήθεια που δίνουν αυτοί μπορεί να αναγνωριστεί ως επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια. Πάντω, αν κάποια από τη βοήθεια αυτή επανέλθει στον προπολογισμό τη ανεπτυγμένη χώρα, τότε αφαιρείται. Τα χρήματα αυτά επενδύονται και επανεπενδύονται στην ανάπτυξη. Και θεωρηθούν αναπτυξιακή βοήθεια, τη στιγμή θα φτάσουν στον κατάλληλο ε, οργανισμό. Η Γαλλία, για παράδειγμα, δεν έχει το σύστημα αυτό, έχει άλλα συστήματα για την χρηματοδότηση της ανάπτυξης. Και η ανάμειξή του στον ιδιωτικό τομέα ε, μετρείται πλέον αναπερίπτωση. Κάθε χώρα θεωρεί ότι το σύστημά της υπερτερεί και θέλουν αναγνώριση του δικού του συστήματος. Αλλά εμείς είμαστε γενόδοροι και στην αναγνώριση άλλων συστημάτων. Υπάρχουν δύο διαφορετικοί ε, δρόμοι που οδηγούν στον, στην ίδιο προορισμό. Δεν λέω ότι το νορβηγικό σύστημα είναι υπέρτερο του γαλλικού ή ανάποδα. Μια χαρά είναι και τα δυο. Τέλος, το άλλο σημαντικό το κόστος για την υποδοχή προσφύγων θα θεωρούνταν επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια για να υπάρξει μια γενναιόδορη πολιτική απέναντι στους πρόσφυγες. Τότε όμως το κόστος της υποδοχής των προσφύγων ήταν πολύ περιορισμένο. Ήταν της τάξης του 3% κατά μέσον όρο. Τώρα, χώρες όπως Αυστρία, ε, Ελβετία και άλλες, αλλά και πολλές χώρες μέλη της Ένωσης έχουν φτάσει σε παραπάνω από 20%. Και πέραν των ε, δαπανών για στήριξη χωρών όπως ε, η Ορδανία, Λίβανος, Τουρκία κλπ. Μόνο για το κόστος υποδοχής των προσφύγων στην επικράτειά τους. Θεωρώ ότι αυτό δεν αποτελεί παραβίαση των κανόνων, αλλά δεν βοηθεί και ιδιαίτερα. Προσπαθώ λοιπόν να συμβουλεύσω τις κυβερνήσεις να κρατήσουν το ποσοστό αυτό χαμηλό. Λέει και η βίβλος νομίζω ότι ε, τα πάντα επιτρέπονται, αλλά τα πάντα δεν είναι και χρήσιμα. Έχουν γίνει κάποιες ε, επιτυχημένες κινήσεις για να μειωθούν τα ποσοστά αυτά. Η Σουηδία έχει φτάσει στο 1,4% για την αναπτυξιακή βοήθεια. Τα μισά θα δοθούν για την υποδοχή των προσφύγων ε, στην επικράτεια. Και τα υπόλοιπα ποσά θα πάνε για άλλες χρήσεις. Οι δύο μεγαλύτεροι δωρητές χορηγή βοήθειας, Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο κατέστησαν σαφές ότι δεν θα πάρουν χρήματα κονδύλια από τον προϋπολογισμό τους για την υποδοχή των προσφύγων στις επικρατείες τους. Προσπαθούμε να κρατήσουμε τα ποσοστά αυτά λοιπόν όσο γίνεται πιο χαμηλά. Είναι όμως υψηλά εν τέλει. Δύσκολο να το κατανοήσει κανείς από τη σκοπιά του αναπτυσσόμενου κόσμου. Πρέπει να δούμε λοιπόν τους κανονισμούς και έχουμε αρχίσει μια διαδικασία για να το εξετάσουμε αυτό. Ποτέ δεν θα είναι εύκολο βέβαια να αλλάξει η κατάσταση αυτή εν μέσω της κρίσης, αλλά πρέπει κάπως να γίνουν πιο αυστηρά τα πράγματα. Να εξεταστεί, για παράδειγμα, αυστηρότερα ο ορισμός του πρόσφυγα. Σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, μπορεί κάποιος να αναγνωρίζεται ως πρόσφυγας. Αυτοί λαμβάνουν την άδεια για να παραμείνουν. Αλλά μπορεί όσοι δεν αναγνωρίζονται ως πρόσφυγες σύμφωνα με τα κείμενα των Ηνωμένων Εθνών μπορεί τελικώς να τους επιτραπεί να παραμείνουν για άλλους λόγους. Και πάντως υπάρχουν μεγάλες διαφορές στην διαμόρφωση των δαπανών ανάμεσα στις χώρες μέλη. Ορισμένα, ορισμένες χώρες της Ένωσης καταβάλουν πολύ μεγαλύτερα ποσά, άλλες πολύ μικρότερα ποσά για τα ίδια θέματα. Οι διαφορές είναι πολύ μεγάλες. Το εξετάζουμε λοιπόν αυτό. Δεν θα είναι εύκολη η πορεία. Θα δούμε ωστόσο αν μπορούμε να εξομαλύνουμε την ε, ε, μορφή αυτή αυτών των διαδικασιών. Αυτά λοιπόν, σας ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε. Ευχαρίστω, είμαι στη διάθεσή για συζήτηση. Σας ευχαριστώ. Μας δώσατε μία πληρέστατη ε, έποψη της κατάστασης. Θα περάσουμε και ωραίο Σαββατοκύριακο. Μας δώσατε έτσι λόγους να είμαστε χαρούμενοι, διότι χθε ο Επίτροπος Λιανίδης ουσιαστικά μας παρουσίασε μια λυσίδα παγκόσμιων καταστροφών. Ξηρασία, Ελληνίνιο, ταξιδεύει από εδώ και από εκεί, αντιμετωπίζει δύσκολες ε, περιπτώσεις, οπότε φαντάζομαι ότι κάποιες φορές νιώθει ότι ο κόσμος γίνεται χειρότερος. Εσείς όμως πολύ σωστά λέτε ότι αν το δούμε στατιστικά, ο μέσος άνθρωπος ε, σε μέσο όρο στις χώρες πηγαίνει καλύτερα, ζει καλύτερα. Στη δική μου ε, τη χώρα σε σχέση με τους ε, γονείς μου από τα 30 ε, όταν δεν υπήρχαν υπηρεσίες υγείας και τα λοιπά σίγουρα η κατάσταση και η δική μου ζωή είναι πολύ καλύτερη. Είναι σημαντικό να θυμόμαστε και το είπαμε ότι χώρες, χώρες όπως είναι σκανδιναβικές χώρες, Γερμανία, ε, και Ηνωμένο Βασίλειο ε, έθεσαν ψηλά τον πύχη όχι όταν είχαν ε, πλουτίσει σαν χώρε, αλλά όταν ήταν φτωχέ. Παραδείγματο χάρη για την υγειονομική υπέρθαλψη κτλ. Και αυτό πρέπει να το έχουμε υπόψη. Και αυτό που είπατε για τι μεταρρυθμίσει, Ήταν σημαντικό να ακούσουμε τη δική σα προοπτική. Ας σας κάνω εγώ τώρα το πρώτο ερώτημα και θα δώσω μετά το λόγο στους συναδέλφους. Το πρώτο ερώτημα λοιπόν είναι Εντάξει, ήσασταν πολύ αισιόδοξο. Είπατε ότι θα πρέπει να δράξουμε την ευκαιρία ε, για να φέρουμε αποτελέσματα. Όμως ε, και άλλες εκθέσεις έχουμε συντάξει, έχουμε πει ότι πρέπει να γίνει κάτι και μετά, μετά από πέντε χρόνια δεν έχει γίνει τίποτα και ξανά από την αρχή και δεν αλλάζει τίποτα. Πιστεύετε εσείς ε, όσα βλέπει κάποια σημάδια πολιτικής βούλησης και αν ναι, πώς μπορούμε εμείς να κρίνουμε ότι κάτι αλλάζει τι θα προκύψει από τον όσα, σε τι ε, θα δεσμευτούν ε, και τι αποτελέσματα θα έχουμε. Το έλκο κύριο Στίαρε έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω τον κύριο Ζολχάιμ. Πρώτα απ' όλα γιατί μας εξήγησε πολύ ξεκάθαρα τις αλλαγές σε σχέση με τη χρήση των ε, στρατιωτικών ε, δυνατοτήτων και μέσων υπήρχε σύγχυση. Τα είπατε πολύ ξεκάθαρα. Με δικά μου λόγια, αν μια αποστολή έχει στρατιωτικού σκοπού, δεν είναι αναπτυξιακή βοήθεια. Αν μπορεί να χρησιμοποιήσει για αναπτυξιακού στόχου κάποια ε, στρατιωτικά μέσα, τότε μπορεί να είναι αναπτυξιακή βοήθεια. Κάπω έτσι είναι τα πράγματα. Αυτή είναι η φιλοσοφία τουλάχιστον η δική σας. Εμείς από πλευράς ΕΛΚ το θεωρούμε θετικό. Υπάρχει και ένα άλλο θέμα. Πέρυσι, στην αναπτυξιακό, στο αναπτυξιακό θεματολόγιο μπήκαν τα ζητήματα ε, της ειρήνης και της ασφάλειας που μέχρι τότε ήταν εκτός. Και ιδίω ε, με τους στόχους ε, βιώσιμης ανάπτυξης για το 2016 μπήκαν και θα πρέπει να δούμε βέβαια και πώς χρηματοδοτείται αυτή το αναπτυξιακό θεματολόγιο. Στα συμπέρασματά σας μιλάτε για την αναθεώρηση της ποσόστοσης σε ό,τι αφορά αποστολές του ΟΗΕ. Ε, είναι σε εξέλιξη φαντάζομαι αυτή η ανάλυση. Διορθώστε με αν κάνω λάθος. Εμείς από τη δική μας πλευρά θα θέλαμε να προχωρήσει κάτι τέτοιο από άλλη από άλλες ίσως ε, πλευρές ε, τα σχόλια να είναι διαφορετικά, αλλά κάπου θα βρούμε φαντάζομαι το συμβιβασμό, τη χρυσή τομή. Θα με ενδιαφέρει όμως να ακούσω από εσάς πού βρισκόμαστε και τι περιμένουμε στο μέλλον. Ευχαριστώ. Έλλη Σλάιν τώρα από τους σοσιαλιστές. Ευχαριστώ. Περιμένω να βάλετε τα ακουστικά. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Σολάιμα. Σε σχέση με αυτό που είπατε στο τέλος της παρεμβασής σας, προφανώς ανησυχούμε. Ανησυχούμε διότι βλέπουμε ότι υπάρχει μία αναδυόμενη τάση να υπολογίζονται οι δαπάνες υποδοχής προσφυγών, προσφύγων με συγχωρείτε, μέλος της ε, επίσημης συναπτυξιακής βοήθειας και παράλληλα βλέπουμε ότι θέλουμε να εγκρίνουμε ένα φιλόδοξο αναπτυξιακό θεματολόγιο με ορίζοντα το 2030. Εγώ νομίζω ότι για να πετύχουμε το θεματολόγιο αυτό χρειαζόμαστε μια καλύτερη δέσμευση από τα κράτη-μέλη, περισσότερους πόρους για την αναπτυξιακή βοήθεια. Ξέρετε ότι η δήλωση της Άντι Σαμπέπα εν μέρη χάθηκε, δεν ολοκληρώθηκε τελικά ως στόχος, διότι δεν υπήρχε απαραίτητη δέσμευση των κρατών που την υπέγραψαν. Επομένως, εσείς μπορείτε να μας διαφωτίσετε λίγο περισσότερο, να μας πείτε τι γίνεται με το Addis Tax Initiative, την φορολογική πρωτοβουλία της Addis Abeba, ζήτημα το οποίο συζητήσαμε και πριν από λίγο με τον πρόεδρο Μπέκη. Νομίζω ότι περισσότερες προσπάθειες πρέπει να καταβάλουμε για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, ιδίω στις συναπτυσσόμενες χώρες. Ποια είναι λοιπόν η δική σας η άποψη σε σχέση με την ε, υποβολή εκθέσεων χώρα, το country by country reporting, πρόταση δηλαδή και πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Νομίζω ότι πρόκειται για μια παγκόσμια πρόκληση την οποία πρέπει να αντιμετωπίσουμε παγκόσμια μέσα. Και συνεπώς δεν μπορούμε να έχουμε μόνο συλλογικά ενοποιημένα δεδομένα στον αφορά τις αμπτυσσόμενες χώρες. Αν πραγματικά θέλουμε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί, θέλουμε πλήρης πληροφορίες, πλήρη ανταλλαγή πληροφοριών ανά χώρα, προκειμένου να δούμε ποια είναι η δράση της κάθε χώρας ξεχωριστά. Η κυρία Χάουτα έχει το λόγο. Σε ευχαριστώ πολύ, Έρικ, για την σφαιρική αυτή εικόνα που μας έδωσες. Είσαι πραγματικά ο κατάλληλο άνθρωπο, κάθε φορά που πρέπει να έχουμε μια σφαιρική εικόνα των πραγμάτων. Ζούμε όμω όντω σε ένα παγκοσμιοποιημένο κόσμο, ο οποίο πολλέ φορέ ομοιάζει με ζούγκλα. Και πρέπει όλοι να συνεχίσουμε να καταβάλουμε προσπάθειες, να συνεχίσουμε να προωθούμε την αναπτυξιακή βοήθεια, να μην χάνουμε τι ευκαιρίε που μα δίνονται μέσω των Panama Papers. Σε σχέση με την πρόσφατη συνεδρίαση της ε, Επιτροπή σου του OECD, της ε, Επιτροπής Αμπτυξιακής Βοήθειας. Διαβάζω ότι ε, ο ΣΑ προσπαθεί να διερευνήσει λίγο περισσότερο πώς χρησιμοποίησε ή πώς ανέφερε την επίσημη αναπτυξιακή της βοήθεια η Δανία, ιδίως όσον αφορά τα προγράμματα εκμάθησης γλωσσών και βοήθειας αναζήτησης απασχόλησης για τους ετούντες άσυλο ενδεχομένως ασφαλμένα να έχει καταχωρηθεί η δαπάνη αυτή ως αντιξιακή βοήθεια. Εσύ μας λες ότι θα πρέπει να παραμείνει χαμηλό το κόστος αυτό. Αρκεί όμως η έκκληση αυτή. Ποιους μηχανισμούς θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε προκειμένου να μην εκτιναθεί το κόστος αυτός, γιατί κινδυνεύουμε πραγματικά αυτή τη στιγμή να καταλήξουμε σε μια τέτοια κατάσταση και να χρειαστεί να πάρουμε πόρους και από άλλους ε, τομείς πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα βαθύτερα αίτια της φτώχειας, για παράδειγμα, που συμβάλλει στη μετανάστευση. Προφανώς εσύ ε, παρακολουθείς πολύ προσεκτικά τα αποτελέσματα και τις συνέπειες της συνδιάσκεψης του, του Μπούσαν για την αποτελεσματικότητα της αναπτυξιακής βοήθειας. Ως προς αυτό τι μπορείς να μας πεις, πόσο πιο αποτελεσματικοί έχουμε γίνει, έχουμε περισσότερους τελικά δωρητές τι γίνεται με αυτές τις νέες μορφές ε, τριγωνικών επαφών και συνεργασίας South-South μεταξύ των χωρών του Νοτίου ημισφαιρίου. Ποιες εξελίξεις βλέπεις εσύ σε αυτό το τομέα. Σάρλ Γκέρλενς από τους Φιλελευθέρους. Ευχαριστώ. Δεν ήμουν και στο εκ των προτέρων συγγνώμη στην εισαγωγή του κυρίου Ζολχάιν, διότι συμμετείχα στη διαπραγμάτευση ενός ψηφίσματος για τις παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου. Πάντως, αν κατάλαβα καλά και ένα θέμα που με απασχολεί και το παρακολουθώ είναι η επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια, σε ποιον δίνεται και ότι κυρίως βέβαια θα πρέπει να προσέξουμε τις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες. Μάλιστα. Πολύ καλά όλα αυτά. Εμείς έχουμε δεχτεί την πρόταση της Κομισιόν για την ε, θέσπιση της αρχής της διαφοροποίησης που εξαιρεί κάποιους δικαιούχους ε, της επίσημης ανάπτυξης βοήθειας από τις ε, χώρες Ένωσης και τις αναδυόμενες χώρες. Αν δει κανεί όμως ότι εκεί υπάρχουν περισσότεροι φτωχοί συμπολίτες μας, τελικά Έχουμε κάποιες ε, αιτιολογίες, για, κάποιες ότι θα πρέπει να λάβουν τις δικές τους ευθύνες αυτές οι αναδυόμενες χώρες εφόσον έχουν έσοδα και θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν την εξαθλίωση του πληθυσμού. Αλλά θα πρέπει αυτές τις ευθύνες να τις συζητήσουν. Δεν έχουμε δικαίωμα παρέμβασης σε αυτές τις χώρες. Όλοι όμως στη μεγάλη διάσκεψη του 2015, νομίζω, προσυπογράψαμε τις αρχές και τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης. Και αυτό συνιστά πρόσκληση προς όλες τις χώρες να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Πώς θα εξασφαλίσουμε την παρακολούθηση αυτών των δεσμεύσεων όσα δεν είναι σε καλή θέση για να προωθεί την ιδέα αυτή του να αναλάβουν περισσότερη ευθύνη τα κράτη-μέλη, γιατί εμείς οι εκτός δεν έχουμε τη δυνατότητα. Πώς μπορούμε να ενεργοποιήσουμε λοιπόν αυτή την ευθύνη ε, των πολύπων. Αυτό είναι το βασικό μου ερώτημα. Ε, κατά δεύτερον, είπατε ότι ένα σημαντικό τμήμα, νομίζω αν μου τα είπαν καλά, είναι ένα 20% της ε, Αναπτυξής Ένωσης, θα μπορούσε ή ίσως ήδη διατίθεται για την μεταχείριση των προσφύγων. Ξέρουμε ποιοι είναι οι προπολογισμοί ε, που δίνουν τα κράτη-μέλη. Δεν ξέρω αν θα είναι αύριο αυτό μια λύση στην κρίση του χρέους που στην Αφρική ε, ανεβαίνει και όταν διαγραφεί, παραγραφεί το χρέος αυτό θα οδηγήσει ε, σε δυνατότητα, ε, θα είναι επιλέξιμες δηλαδή αυτές οι χώρες για να λάβουν επίσημα αναπτυξιακή βοήθεια. Άρα τελικά υπολείπεται σημαντικά η βοήθεια που πραγματικά δίνεται σε σχέση με αυτό που φαίνεται ψήμως. Πριν καμιά δεκαπενταρία χρόνια είχα διαβάσει στην εφημερίδα Le Monde ένα άρθρο για τον ΟΣΑ με τίτλο να είστε λίγο πιο, λιγότερο διακριτικοί, παρακαλώ. Εγώ θα σας ζητήσω να είστε εντελώς αδιάκριτοι και αν δεχτείτε και το κάνετε τελικά, νομίζω ότι θα έχετε και την πλήρη υποστήριξή μας. Άρα να είστε και πιο τολμηροί από ό,τι ε, είσαστε μέχρι τώρα. Κύριε Ζολχάιμ, έχετε το λόγο πάρα πολύ καλές ερωτήσεις και πολλές στον αριθμό. Σας το προκαταβολικά, συγγνώμη, είτε αν δεν απαντήσω σε όλες, είτε αν δεν δώσω πλήρης απαντή σε όλες τις ερωτήσεις σας. Να ξεκινήσω από τον ε, τελευταίο μιλητή. Όχι, δεν μιλάω για το 20%. Σε κάποια κράτη-μέλη, δεν μιλούσα για το σύνολο των προσφύγων. Και ξέρω Γερμανία και Ηνωμένο Βασίλειο, τους δύο μεγαλύτερους δωρητές. Και βέβαια η ΙΠΑ, η Ιαπωνία και άλλες χώρες δεν ε, αφορούνται. Άρα μιλάμε για ένα πολύ πιο σημαντικό τμήμα. 20% όμως σε κάποιες χώρες, σκανδιναβικές για παράδειγμα. Δεν είμαι απόλυτα βέβαιος, αλλά νομίζω το ίδιο ισχύει για Αυστρία, Ελβετία και Ολλανδία. Αλλά σε περισσότερες χώρες πολύ χαμηλότερο το ποσοστό. Μέχρι τώρα στη ζωή μου κατέληξα στο συμπέρασμα ότι ο σημαντικότερος παράγοντας για την παρακολουθία είναι η ηγεσία και αυτό βέβαια είναι το σημαντικότερο παντού και για την Ευρώπη και για οποιαδήποτε άλλη χώρα και για οποιοδήποτε τομέα. Μπορεί να είναι δύο κράτη παρόμοια σε πολλά και να έχουν τεράστιες διαφορές στην ανάπτυξη. Βόρεια Νότια Κορέα για παράδειγμα. Αλλά Ερυθρέα Αιθιοπία είναι ένα άλλο παράδειγμα. Γιατί η Ερυθρέα μένει πίσω και η Αιθιοπία προχωρά. Ή δείτε, Αιτή, η Δομινικανή Δημοκρατία. Η Δομινικανή Δημοκρατία είναι 7 φορές ε, ε, πλουσιότερη, κατά κεφαλήν μιλάω, σε σχέση με την Αιτή. Άρα δεν έχουν όλα να κάνουν με την ηγεσία. Δεν είναι τέλειοι σίγουρα, αλλά σε κάποιε χώρες όπως στη Δομινικανή Δημοκρατία δεν είναι δικτάτορε ή τόσο ηλίθιοι όπως είναι στην Αϊτή. Και το θέμα είναι να επηρεάζει η ηγεσία τελικά. Για την Χάιντι Χάουταλ που μίλησε για τη διάσκεψη του Μπουσάν. Δυσκολευόμαστε. Ιδίως ό,τι αφορά τη δημοσιονομική στήριξη που ήταν από τα πορίσματα του Μπουσάν είναι κάτι που από πολιτική πλευρά ε, αποδείχθηκε πάρα πολύ δύσκολο. Πρέπει να σα απασχολήσει και εσά. Υπάρχουν και άλλε πολιτικέ δυσκολίε που αντιμετωπίζουν βέβαια οι Ευρωπαίοι πολιτικοί. Και να σα πω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Παρέχεται δημοσιονομική υποστήριξη στην Ουγγάντα. Και έπειτα ο πρόεδρο Μουσέβη παρουσιάζει για του ομοφυλοφίλου ένα νομοσχέδιο που η κοινή γνώμη στην Ευρώπη το κατακρίνει. Και είναι πάρα πολύ δύσκολο να συνεχιστεί αυτή η δημοσιονομική υποστήριξη και επιλέγεται κάτι διαφορετικό για την κοινωνία των πολιτών, τα μέσα μέσα ενημέρωση η αντιπολίτευση στο κοινοβούλιο θα ζητήσει να υπάρξει αντίδραση αφού μπορεί απ' την άλλη να είναι τελείως διαφορετικό το τι πιστεύει η η γνώμη στην Ουγγάντα από τι πιστεύει η Ευρωπαϊκή Ένωση για τους ομοφιλόφιλους. Δεν σας ακούω. Είναι κληρονομιά της αυτοκρατορίας, ξέρετε, η νομοθεσία στην Ουγγάντα. Ναι, πράγματι, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι είναι δύσκολο να υποστηριχθεί από τους ευρωπαίους πολιτικούς η δημοσιονομική υποστήριξη όταν η κοινωνία των πολιτών, τα μίντια και άλλοι ασκούν κριτική ε, σε ένα αναψώμενο κράτος για κάποια πολιτική του. Οπότε περνάνε σε κάποιο άλλο μέσο. Δεν μπορώ να το λύσω εγώ αυτό. Νομίζω ότι μπορείτε να το συζητήσετε εσεί μεταξύ σα. Αλλά αν θέλετε πραγματικά να δώσετε δημοσιονομική υποστήριξη, θα πρέπει να είστε λίγο πιο αποφασιστικοί απέναντι σε κάποιε αρνητικέ στάσει. Η συνεργασία νότου-νότου πράγματι αυξάνεται. 130 δις νομίζω σε δολάρια, άρα και σε ευρώ κάπου αντίστοιχο είναι το ποσό με βάση τις αλλαγματικές ισοτιμίες και τα λοιπά, αλλά αν προσθέσετε Κίνα και τους Άραβες, αυξάνεται πολύ αυτό το πόσο. Η Κίνα συνεισφέρει περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο στην συνεργασία νότου-νότου. Και άλλοι όμως. Αν έχουμε μια μικρή ομάδα που δίνουν και όπως η και μια μικρή ομάδα που, που δέχονται όπως το Μαλάου, θα πρέπει να δούμε τι γίνεται. Η χιλή, να σας δώσω ένα παράδειγμα. Θα γίνει σύντομα μια χώρα υψηλού εισοδήματο αντί για χώρα μεσίου εισοδήματο. Θέλουν όμως να παραμείνουν αποδέκτες της βοήθειας. Γιατί λένε η Παραγουάη που δεν τα έχει καταφέρει τόσο καλά, είναι πιο ατυχής έχει τη βοήθεια, αλλά θέλουν να πάρουν βοήθεια και οι χιλιανοί. Γιατί λένε ότι δεν μπορούμε αλλιώ να εφαρμόσουμε τους ε, στόχους βιωσιμότητα και να τηρήσουμε τα συμπεφωνημένα στο θεματόλογο 2030. Αυτά λοιπόν τα νέα ζητήματα που θα πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε. πρέπει να δούμε σε ένα είδος ισολογισμού τι γίνεται με την παροχή βοήθειας και την υποδοχή της βοήθειας. Υπάρχουν πολλές προκλήσεις ακόμη. Ε, δεν μπορώ να σχολιάσω δηλαδή, τα δημοσιεύματα του οποία τη Δανία. Τα περισσότερα κράτη νομίμως, νομίζω, αξιοποιούν αυτές τις σχέσεις. Αν υπάρχουν καταχρήσεις, θα το δούμε και θα το καταγγείλουμε. Δεν μπορώ να σας πω τι γίνεται με τη Δανία. Θα το εξετάσουμε πάντως σε επίπεδο ΩΣΑ. Για την κυρία Σλάιν. Πρέπει να υπάρχει πλήρης διαφάνεια στις διεθνείς κεφαλαϊκές ροές. Πώς μπορούμε να δεχθούμε να υπάρχει διαφάνεια σε όλους τους άλλους τομείς. Αφού υπάρχει και απαιτούμε διαφάνεια παντού και θέλουμε να λαμβάνονται και οι πολιτικές αποφάσεις με διαφάνεια, πώς μπορούμε να δεχθούμε να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Τη δεκαετία του 90 είχαμε μια τραγωδία θαλάσσια. 150 άτομα έχασαν τη ζωή τους ε, ε ψακτές Κοπενχάγης, ε, έπιασε φωτιά σε ένα πλοίο. Και Παρότι έχουν περάσει πάνω από 25 χρόνια από τότε, δεν ξέρουμε ακόμη τι έγινε που οφείλεται η τραγωδία αυτή. Όλα ήταν στο κυβερνοχώρο. Τελικά δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε τι έγινε. Παρ' αυτά, παρότι έχουμε τη δυνατότητα, δεν καταφέραμε. Πώς θα το καταφέρει τον Νεπάλι το Καμερούν. Θέλουμε να έχουμε ένα πιο υπεύθυνο καπιταλισμό. Πώς θα γίνει αυτό, αν δεν γνωρίζουμε τον ιδιοκτήτη ενός εργοστασίου ή τον κάτοχο μεγάλων σημαντικών ποσών. Άρα η εκθέση αναχώρα, η εκθέση αναχώρα εκθεση πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο, θα το στηρίξουμε, θέλουμε να γίνει πράξη και όχι μόνο εντό Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά φυσικά και για του φορολογικού παραδείσου και του άλλου προορισμού. Είναι κομβικό. Έχουμε ξεκινήσει και άλλους πρωτοβουλίες, φορολογική πρωτοβουλία για παράδειγμα να βοηθήσουμε τις φορολογικές διοικήσεις των ψωμένων χωρών. Έχουμε τους φορολογικούς επιθεωρητές ε, χωρίς σύνορα για την παροχή τεχνικής ε, ε, εμπειρίας, τεχνογνωσίας. Έχουμε και κάποιες συμφωνίες που κοιτάμε, πάνω χάρη συμφωνίες με τις εξορρεκτικές βιομηχανίες. π.χ. η Σερβία ή η Αυστραλία. Θέλουμε να εξασφαλίζεται σωστός συσχετισμός δυνάμεων. Και προβλεψιμότητα βέβαια χρειάζεται για τις επιχειρήσεις, αλλιώς θα υπάρξουν επενδύσεις. Γι' αυτό θέλουμε να παρέχουμε και την βέλτιστη δυνατή τεχνογνωσία και αναφερθήκαμε και στην πρωτοβουλία αυτή για τη διάβρωση της βάσης και τη μεταβίβαση των κερδών. Αναφίβολα, προφανώς, τα πράγματα έχουν τροποποιηθεί. Θεωρώ ότι έχουμε θετικές εξελίξεις, αλλά θα πρέπει αυτές να επιταχυνθούν. Και δεν μπορούμε να επιταχύνουμε τις θετικές εξελίξεις αν δεν έχουμε την κατάλληλη πολιτική ηγεσία και την κατάλληλη πολιτική πρωτοβουλία. Μετά την οικονομική κρίση είδατε ότι οι Υπουργοί Οικονομικών από τις περισσότερες αναπτυγμένες χώρες και με τη βοήθεια, με τη βοήθεια των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και με χώρες όπως η Βραζιλία και η Ινδία είπαν ότι δεν μπορούμε πλέον να έχουμε διαφεύγοντα κέρδη. Θα πρέπει να συλλέγονται σωστά οι φόροι. Πρέπει να έχουμε τους πόρους αυτούς. Ξαφνικά ανακάλυψαν ότι υπήρχαν τεράστια νομικά κοινά και ότι υπήρχαν πάρα πολλοί εύποροι που μπορούσαν να βγάζουν τα χρήματά τους στο εξωτερικό χωρίς να καταβάλουν καθόλου φόρους. Τα πράγματα αλλάζουν μόνο όταν υπάρχει πολιτική ηγεσία όταν υπάρχει απαραίτητη πολιτική βούληση. Και αυτό βρίσκεται και στην καρδιά του λεγόμενου υπεύθυνου καπιταλισμού. Δεν σας λέω αυτή τη στιγμή κάτι το επαναστατικό. Ο καπιταλισμός θα πρέπει να λειτουργεί όπως είχε σχεδιαστεί να λειτουργεί. Αν λειτουργούσε σωστά το σύστημα, δεν θα υπήρχαν τόσοι πολλοί που να μπορούν να κρύβουν τα χρήματά τους στις Βρετανικές Παρθένες νήσους ή σε άλλα μέρη. Το σύστημα υπάρχει, πρέπει απλώς να λειτουργεί σωστά. Κύριε Στίερ, εσείς αναφέρατε δύο ακόμα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ειρήνη και την ασφάλεια. Α μην εθελοτυφλούμε εδώ πέρα. Όντω, τα δύο αυτά ζητήματα είναι πάρα πολύ σημαντικά για την ανάπτυξη. Αν οι Γάλλοι δεν είχαν επέμβει στην κεντροαφρικανική δημοκρατία, θα είχαμε μια τεράστια καταστροφή στη χώρα αυτή. Και καταλαβαίνετε ότι αυτό θα είχε πειράσει πάρα πολύ αρνητικά και τη χώρα αυτή και τις γύρω περιοχές αν οι Γάλλοι δεν είχαν επένδυση στο Μαλί επίσης, κατά πάση πιθανότητα η χώρα αυτή, εν μέρη τουλάχιστον, θα είχε καταληφθεί από τζιχαντιστές. Καταλαβαίνετε λοιπόν και η παρέμβασή τους ήταν καθοριστική. Δεν μπορούμε όμως να χρηματοδοτούμε τις στρατιωτικές παρεμβάσεις μέσω της επίσημης ναπτυξής βοήθειας γιατί θα πάρουμε κατά αυτόν τον τρόπο χρήματα από άλλους τομείς όπως η παιδεία και η εκπαίδευση. Πρέπει λοιπόν να δούμε εδώ τα περιθώρια τα οποία έχουμε. Τέλος, Δέκα χρόνια από τη ζωή μου ασχολήθηκα με διάφορες ειρηνευτικές διαδικασίες, όπως στη Σρι Λάγκα. Νομίζω ότι πετυχαίνουμε την ειρήνη μόνο όταν έχουμε τις σωστές πολιτικές. Μπορείτε να βοηθήσετε αποσπασματικά μέσω χρημάτων, μπορείτε να επέμβετε και με στρατό, αλλά αν δεν καταφέρετε αργά ή γρήγορα να, να καταλήξετε στις σωστές πολιτικές, ε, δεν πετυχαίνετε ποτέ μια βιώσιμη ειρήνη όπου είχαμε ημίμετρα στο παρελθόν, όπου δεν είχαμε δηλαδή τις σωστές πολιτικές, δεν καταφέραμε να καταλήξουμε σε μία μόνιμη βιώσιμη ειρήνη. Πρέπει λοιπόν να καταφέρουμε να βελτιώσουμε και εκεί τις επιδόσεις μας, αλλά και στον τομέα αυτό της ειρήνης και της ασφάλειας, πάλι τα πηγαίνουμε καλύτερα σε σχέση με το παρελθόν. Βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή έχουμε αναπτυσσόμενες χώρες, όπως η Τανζανία, οι οποίες από πολιτικής πλευράς τα πηγαίνουν καλύτερα από ότι άλλες χώρες που βρίσκονται σε πιο κρίσιμη πολιτική κατάσταση, όπως το Νότιο Σουδάν. Επί του παρόντος, στο Νότιο Σουδάν, ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος ακόμα αντιμάχονται μεταξύ τους σε σχέση με διάφορες ε, πολιτικές που πρέπει να εγκριθούν, ενώ παράλληλα πάρα πολλοί άνθρωποι σε καθημερινή βάση στη χώρα αυτή χάνουν τη ζωή τους. Καλούμεθα λοιπόν εμείς να θεραπεύσουμε την κρίση αυτή, καλούμεθα να ενισχύσουμε την ανθρωπιστική μας υποστήριξη στη χώρα αυτή, ενώ βλέπουμε ότι παράλληλα δεν υπάρχει καμία διαφάνεια για το πώς δαπανώνται τα χρήματα τα οποία δίνουμε εμείς στο Νότιο Σουδάν, μια χώρα που συνεχίζει να πλήττεται από τον πόλεμο, ένας πόλεμος που σκοτώνει πολλούς ανθρώπους και καθιστά πλούσιους και ακόμα πλουσιότερους κάποιους άλλους. Νομίζω λοιπόν ότι ακριβώς τέτοιες καταστάσεις θα πρέπει να αποφύγουμε. Αυτή τη στιγμή θα πληρώνουμε εμείς για την ανθρωπιστική βοήθεια που πηγαίνει σε μια χώρα. Ε, πρέπει παράλληλα να υπάρχει ένα διαφανές καθεστώς στα πλαίσια του οποίου θα βλέπουμε πώς δαπανώνται ακριβώς τα χρήματα. Αυτό θέλουμε να δούμε στο Νότιο Σουδάν. Ποιε επίση είναι οι τράπεζε αυτέ οι οποίε στην Ευρώπη και σε άλλε περιοχέ του αναπτυγμένου κόσμου παίρνουν χρήματα αυτή τη στιγμή από τον Νότιο Σουδάν. Τι κάνουν με τα χρήματα αυτά. Και αυτά πρέπει να παρακολουθούμε, λέει η Πρόεδρο. Πρέπει να δούμε ποιοι τραπεζικοί λογαριασμοί υπάρχουν με χρήματα τα οποία έχουν διαφύγει από τον Νότιο Σουδάν και που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν με έναν πολύ διαφορετικό τρόπο. Ο Έρικ πάντως για άλλη μια φορά μας έδωσε πολύ τροφή για συζήτηση. Προφανώς θέλουμε να συνεργαστούμε και μαζί σας και με τον Τάμπο Μπέκη. Καταγράφουμε λοιπόν όλες αυτές τις πληροφορίες που μας δώσατε. Έχουμε όμως και εκπροσώπους από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο Ζεγόμ Λεγουά ενδεχομένω. Θέλετε λίγο να μας διαφωτίσετε για τη σχετική δράση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ Πρόεδρε, θα προσπαθήσω να είμαι πάρα πολύ σύντομος. Δύο λεπτά μόνο θα μιλήσω. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμμετέχει ενεργά στην διαδικασία επανοργάνωσης της επίσημης συναπτυξιακής βοήθειας και μάλιστα συμμετέχουμε και στην Επιτροπή Αναπτυξιακή Βοήθειας του ΟΣΑ. Όντω, η εικόνα που μα δώσατε είναι ιδιαίτερα σφαιρική και αντιπροσωπευτική. Είμαστε υπέρ τη πρωτοβουλία τη φορολογική τη Αντίσα Μπέπα. Θεωρούμε ότι θα πρέπει να έχουμε μια ολιστική προσέγγιση που να περιλαμβάνει το σύνολο τη διαχείρισης των δημοσίων δαπανών όχι μόνο τα έσοδα τα οποία προέρχονται από τη φορολογία, αλλά και τα υπόλοιπα έσοδα τα οποία καλείται να συλλέγει ένα κράτο. Όσον αφορά την ειρήνη και την ασφάλεια, είμαστε υπέρ τη μικρή αυτή μεταρρύθμιση που κάνετε. Συμμετείχαμε και εμεί στην όλη διαπραγματευτική διαδικασία όσον αφορά τα δάνεια. Σημαντική γίνεται η προσπάθεια που γίνεται εδώ πέρα. Τα δάνεια αποτελούν σημαντικό τμήμα τη γενικότερη εργαλειοθήκη που έχουμε. Η εν εξελίξει μεταρρύθμιση είναι ικανοποιητική, συμφωνούμε με τις προτάσεις γραμματείας και με τις τελευταίες προτάσεις που έχουν να κάνουν με τα μέσα του ιδιωτικού τομέα. Για πολλούς όμως λόγους ε, είμαστε περισσότερο υπέρ μιας ε, προσέγγισης που χρησιμοποιεί περισσότερα εργαλεία τεχνικά και όχι τόσο πολύ θεσμικά εργαλεία. Θεωρούμε ότι ε, τα τεχνικά μέσα μας δίνουν μεγαλύτερη ακρίβεια και μεγαλύτερη διαφάνεια. Ωστόσο, είμαστε ικανοποιημένοι και με την υφιστάμενη κατάσταση και ελπίζουμε ότι το 2016 θα καταφέρουμε να ολοκληρώσουμε το πρόγραμμα αυτό προκειμένου να μπορέσουμε να το εφαρμόσουμε το συντομότερο δυνατό μετά. Τώρα, όσον αφορά το κόστος υποδοχής προσφύγων σε μια χώρα. Νομίζω ότι πρέπει να ευθυγραμμιστεί ο τρόπος ε, καταμέτρησης των δαπανών αυτών. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι τα μέλη της ΔΑΚ χρησιμοποιούν εντελώ διαφορετικές μεθόδους καταμέτρησης αυτών των δαπανών. Και αν δεν κάνω λάθος έχετε δημιουργήσει μια ομάδα εργασία η οποία θα επιληφθεί του ζητήματος. Αυτό μας ικανοποιεί ιδιαιτέρως. Τέλος, κάτι το οποίο δεν έφερε ο κύριος Σοντχάιμ είναι το TOSSD, συνολική επίσημη υποστήριξη για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Το ODA, η επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια, αποτελεί ένα μόνο μέρος των κεφαλακών αυτών ροών. Εσείς αυτή τη στιγμή δημιουργήσατε ένα νέο μέσο, τη συνολική επίσημη υποστήριξη για τη βιώσιμη ανάπτυξη, το TOSSD, Αυτά τα νέα συνολικά αριθμητικά δεδομένα λοιπόν θα είναι ιδιαίτερα χρήσιμα όσον αφορά τη στατιστική μας ανάλυση και θα ήθελα να ζητήσω και από τον ΟΣΑ να αρχίσει να χρησιμοποιήσει το νέο αυτό στατιστικό μέσο το συντομότερο δυνατό προκειμένου μέσα σε ένα 1,5 χρόνο να έχουμε θετικά αποτελέσματα. Μα δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω με όλα αυτά τα οποία είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Πρόεδρος, μα και ο Επίτροπος ε, Μέμιτς προκείται να έρθει στα πλαίσια του διαρθρωμένου διαλόγου. Ενδεχομένως ε, θα μπορούσαμε από τον ε, Επίτροπο, τον κύριο Μίμητσα, να το πούμε τι κάνει ο ίδιος στο δικό του χαρτοφυλάκιο, τι κάνει όμως και το σύνολο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Για παράδειγμα, τι κάνει και η κυρία Μογκερίνη στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της. Ας μην ξεχνάμε ότι στα πλαίσια των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης καλύπτουμε ουσιαστικά τις περισσότερες από τις αρμοδιότητες των επιτρόπων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πρέπει λοιπόν να καταφέρουμε να δούμε τι κάνουν οι επίτροποι και τι κάνουν βέβαια και οι υπόλοιπε επιτροπές του Κοινοβουλίου. Έρικ, για άλλη μια φορά σε ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σου εδώ σήμερα. Δεν μπορούμε να καλύψουμε τα άλλα δύο σημεία. Δεν υπήρχαν άλλωστε τίποτα στα διάφορα. 23 Μαΐου είναι η επόμενη συνεδρία, 23 και 24 Μαΐου. Η Πρόεδρος ευχαριστεί και τους διερμηνείς. Σας ευχαριστώ πολύ.